Η Σίτσομ... Επαναλαμβάνεται η συνεδρίαση. Να σας ενημερώσω ότι η έκθεση Λαβία για τον διορθωτικό προπολογισμό 1 κάτω 2013 για τις δαπάνες που σχετίζονται με την ένταξη της Κροατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και η έκθεση Μπέγκερ για την τροποποίηση της Διοργανικής Συμφωνίας της 17ης Μαΐου 2006 για τη Δημοσιονομική Πειθαρχία για να ληφθεί υπόψη η ένταξη της Κροατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ιδιαίτερα οι δαπάνε προκύπτουν από αυτό, αυτές οι δύο εκθέσει αποσύρθηκαν από την ημερήσια διάταξη. Στην Δευτέρα, 10 Ιανουαρίου 2013, ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου εξήγησε την ουσία της κατάστασης. Επειδή δεν ήταν σε θέση το Συμβούλιο να στείλει το, την θέση του στο Κοινοβούλιο, δεν μπορούμε για αυτά τα σημαντικά θέματα να πάρουμε θέση αυτή τη βδομάδα. Να περάσουμε τώρα στις προφορίε. Να αρχίσουμε με βάση την ε, απλοποιημένη διαδικασία άρθρο 138 του κανονισμού για την έκθεση του κυρίου David Μάρτιν για την ενδιάμεση συμφωνία εταιρική σχέσης Ευρωπαϊκής Ένωσης και Κεντρικής Αφρικής. Να ψηφίσουμε. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά.